του Κοινοβουλίου απολάβουν όλων των δικαιωμάτων ε, όμως θα πρέπει πρώτα να έχουν ε, υπογράψει την ε, δήλωση ότι δεν κατέχουν κάποια θέση ασυμβίβαστη. Τώρα, όσον αφορά την συνήθη νομοθετική διαδικασία, σας ενημερώνω ότι την Τρίτη Μαζί με τον πρώτο Συνοβουλίου έχουμε κάποια υπογραφή κάποιων νομοθεμηνών σύμφωνα με την διάταξη 74